witam serdecznie panie i panowie bardzo proszę kto opuszcza salę o opuszczanie po cichu. Σας καλωσορίζω όλους. Παρακαλώ, φεύγουν από την αίθουσα λίγη ισχύα. Ακολουθεί τώρα συζήτηση για την πολιτική ακαιρεότητα της Επιτροπή, ιδίω όσον αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Ο κύριος Έτιγκερ έχει τον λόγο πρώτος. Ο επίτροπο. παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι,